So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Έχουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, συζήτηση με την Βελγική Προεδρία. Σας καλωσορίζω θερμά όλους, ιδιαίτερα την κυρία Σάουφλεγκε, η οποία είναι η εκπρόσωπος της Προεδρίας, Υπουργό Περιβάλλοντος Φύσης και Πολιτισμού και Πρόεδρος του Και ο κύριος Φανπέτριν είναι εδώ, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου. Άρα το Συμβούλιο εκπροσωπείται από τον κύριο Πιέτρας και θα παρακολουθήσει την παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας. το άτυπο συνεδρίαση στη Γάνδη των Υπουργών Περιβάλλοντος ήταν ε, η πρώτη συνεδρίαση που οργάνωσε η Βελγική Προεδρία. Σας συγχαίρω, πρόκειται για μια συζήτηση για την ε, διαχείριση των πόρων στην Ευρώπη χτες και σήμερα. Μάλλον Δευτέρα και Τρίτη. Πρόκειται για ένα τομέα αρκετά ε, αβέβαιο σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί είναι οι τομεί που μας απασχολούν με προτάσεις νομοθετικές που θα δούμε στο μέλλον και πιστεύω ότι θα βρείτε μία λύση για την διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, των βιολογικών αποβλήτων, όπου έχουμε επίσης μία πρόταση Φυσικά θα αναφέρω ακόμη και τη βελτίωση ε, των διατάξεων για τα ελαφρά οχήματα, τα βιοκτώνα, το σχετικό κανονισμό από το χώρο της, της χημίας, όπου επιδιώκεται συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όπως είπα, είναι σημαντικές οι στιγμές που ζούμε τώρα ε, με μία μεγάλη διάσκεψη τον Οκτώβριο για την βιοπικιλότητα και για την προστασία της, από την κλιματική αλλαγή. Και ελπίζουμε οι δυσάρεστες ε, εμπειρίες της Κοπενχάγης και του Αγαδίρ να αποτελέσουν δίδαγμα για την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη. 27 κράτη-μέλη συν την Επιτροπή, 28 δεν σημαίνουν απαραίτητα μια μεγάλη μονάδα. Έχουμε μάθει δυστυχώς ότι όταν δεν μιλούμε όλη την ίδια γλώσσα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη γιατί πρέπει να εκφράζουν όλοι κοινέ θέσει, την ίδια θέση. Και ελπίζω και στο Κανκούν αλλά και στην Αγκόγια να εκφραστεί μία και ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε περιθώρια για άλλα ισχνά αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε θάρρος, χρειαζόμαστε στράτευση. Διαφορετικά τα προβλήματα επιδεινώνονται διαρκώς και λύσεις δεν έρχονται. Βλέπω με χαρά ότι όλοι οι Βέλγοι συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής μας, είναι παρόντες, αλλά ασφαλώς και από τις άλλες πολιτικές ομάδες, πολύ σημαντικοί συνάδελφοι, προσβλέπω σε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί σας και σας δίνω το λόγο για την παρουσίαση. Uh, uh, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας για το Περιβάλλον εδώ ενώπιον της ε, Επιτροπής σας. Και ως ε, Προεδρία εκτιμούμε το έργο το οποίο επιτελείται και την εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη σας όσον αφορά τα θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας τροφίμων. Πάντοτε έχει διδάματι ρόλο όσον αφορά τις εξελίξεις στην πολιτική του περιβάλλον και η Βελική Προεδρία έχει επίγνωση του ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Λισαβόνα έχει έναν ρόλο αναβαθμισμένο στα θέματα του περιβάλλοντος και βέβαια ήδη πριν την σύνδεση της Λισαβόνας είχαμε την ε, διαδικασία της συναπόφασης που ήταν τότε η φυσιολογική νομοθετική διαδικασία οπότε ήδη προϋπήρχε ε, διάλογος μεταξύ ημών και ημών. Έτσι καταφέραμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και για μένα ως φλαμαδής υπουργού για περιβάλλον και πολιτιστικά. Είναι τιμή να σας παρουσιάζω ένα τέτοιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα για το περιβάλλον, το οποίο είναι πρόγραμμα κλειδί για την Προεδρία μας. Έχει πολλές προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αυτή την πάρα πολύ χειρότερη κρίση εδώ και μισό αιώνα. Προβλήματα με απασχόληση και κοινωνική πολιτική. Επίση, το αρμοδοπιστωτικό σύστημα και η ανταγωνιστικότητα έχουν πληγεί. η, αυξάνεται ο πληθυσμό τη γη, αυτό σημαίνει πίεση για το περιβάλλον, οπότε επιβάλλεται μια εκβάθρον αναδιοργάνωση τη οικονομία και του περιβάλλοντο. Και, και ε, έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε πρωταγωνιστέ στη δημόσια σκηνή. Ε, έχουμε τώρα κάποιες ε, άλλες προκλήσεις. Έχουμε το στόχο της ε, οικονομίας με λίγη χρήση άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα οπότε θέλουμε προς τα κύριο της Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕ Προεδρία έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένο και μπορούμε να το υλοποιήσουμε αν ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαστούμε συνδυάσουμε τις δύναμεις μας και έτσι στείλουμε ένα κοινό μήνυμα Οπότε θα υπολογίσουμε και εμεί τη βοήθειά σα να σα πω τώρα τις προτεραιότητες μας, τις προτεραιότητες της που είναι τέσσερι. Ξεκινώ με το θέμα του κλίματος. Μετά την Κοπενχάγη πρόκειται να έχουμε την διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην Κανκούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε ότι έτσι θα ανακτήσουμε εμπιστοσύνη. Ε, ελπίζουμε ότι ε, θα μπορέσει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Προεδρία και δεν θα υστερήσει. Και χθε στην Γάνδη είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων. Όλα τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση βαθμιαία με μικρά βήματα να πάμε στην Κανκούν και να προσπαθήσουμε να πείσουμε για τις προτάσεις μας τα άλλα τα άλλα κράτη που θα είναι εκεί στην Κανκούν και επίσης να θα με την ανοτεχνολογία, τη μεταφράση τεχνολογίας ε, και το MRV, στα αγγλικά Monitoring Verifying Reporting, παρακολούθηση, εξακρίβωση και ε, αναφορά. Θέλουμε να υπάρξει ένα πλαίσιο όπου να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας και θέλουμε να έχουμε πάνω από 20% των βλαπτικών για το περιβάλλον αερίων. Έχουμε και κάποιες διαρροές του διοξιδίου και θα πρέπει να μελετήσουμε ξανά αυτή την πρόκληση για να δούμε τι θα γίνει με την πρόταση για μείωση 30%. Να δούμε αν αυτό το 30% μπορεί να είναι ρεαλιστικός στόχος. Επίσης, έχουμε συμφωνήσει στην Κοπενχάγη για χαμηλό επίπεδο εκπομπών στις πόλεις μας μέχρι το 2050. Κατά την Ισπανική Προεδρία, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος εξέτασε αυτό το ζήτημα του θα ξαναεξεταστεί στην Συνοδό του Οκτωβρίου. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να επεξεργαστεί τα διαφορετικά σενάρια και πρόκειται να μα αναφέρει σχετικά και να κατεβάσει συγκεκριμένε προτάσει. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, έχετε να το συζητήσει περαιτέρω και που έχετε να βοηθήσει ούτω ώστε να ληφθούν ε, κάποιε αποφάσει τον Οκτώβριο. Επίση, επεξεργαζόμαστε το πώ θα μπορέσουμε να μειώσουμε τι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακο από τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Εάν έχουν οριμάσει τα πράγματα, μπορεί και σε πρώτη ανάγνωση να κλειστεί κάποια συμφωνία επιβελική Προεδρία και αυτό θα είναι πάρα πολύ ευχαριστώ για μα. Δεύτερη προτεραιότητά μα είναι η βιοπικιλότητα. Το 2010, που γνωρίζετε, είναι το Διεθνέ Έτο για την Βιοπικιλότητα. Η δε Προεδρία θα ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευμενή συγκυρία για να μπορέσουμε να σημειώσουμε μια σημαντική πρόοδο. Αυτό μπορεί να γίνει στην ε, συνάντηση την συναγκόγια και έχουμε διάφορους ε, δείκτες που κατατείνουν στο ότι ε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να το προσέχουμε. 15 ε, Μαρτίου συζητήθηκε στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος το τι μπορεί να γίνει βράχη πρόθεσμα όσον αφορά την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Και θέλουμε να πάρουμε και εμείς τη σκητάλη, να συνεχίσουμε το ίδιο θέμα, θέλουμε να συσπυρώσουμε το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη σε μια συνένεση για να υπάρχει ένα θετικό ε, αποτέλεσμα για τους φιλόδοξους στόχους για το στρατηγικό πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2010. Σήμερα ήδη έχουν αρχίσει στο Μόντρεαλ οι συζητήσεις για το τι θα γίνει με το ABS, Access and Benefit Sharing. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μία ενιαία φωνή όπως και στην Αγκόγια. Το ΔΕ Συμβούλιο Περιβάλλοντος το, του Δεκεμβρίου θα λάβει αποφάσεις με αποτέλεσμα τα όσα θα προκύψουν στην Αγκόγια είναι πάρα πολύ σημαντική βιοποικιλότητα για το οικοσύστημα και για την ευημερία μας για το, και για την οικονομία. Ε, υπάρχουν ε, οι υπηρεσίες που σχέση με το περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τα έχετε συζητήσει εδώ πολλές φορές. Έχουμε την έκθεση του tafepson b The Economics και Ecosystems και Biodiversity και οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα και θέλουμε να είναι αηφόρες οι επιλογές σε σχέση με την βιοποικιλότητα και το βιοσύστημα και το οικοσύστημα μάλλον να μην τίθεται εν κινδύνο. Ε, επίσης στη συνέχεια πρόκειται να συζητήσουμε για τα τροποποιημένα και όπως ξέρετε είχε αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία ο κ. Ντάλι που τα συζήτησε μαζί σας χθε. Και στα πλαίσια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος όλα αυτά έχουν συζητηθεί. Η Βελική Πρόεδρε πρόκειται να συνεχίσει αυτή τη συζήτηση ε, στην ίδια γραμμή πλεύση. Τώρα έχουμε την τρίτη μας προτεραιότητα που είναι η διαχείριση των αηφόρων των βιώσιμων υλικών. Είπαμε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει να προσέξουμε τις επικαλύψεις μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Να βρούμε κάποια μέσα και εργαλεία ούτως ώστε να μπορέσουμε ε, και το περιβάλλον και την οικονομία σαν πολιτικές να τις ε, εξελίξουμε. Θέλουμε επίσης να είμαστε αποτελεσματικοί για τις ενέργειες, να έχουμε επομένως μια τέτοια ε, διαχείριση των αηφόρων βιώσιμων υλικών. Αυτό σημαίνει αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση υλικών, φυσικών πόρων αλλά και αποβλήτων θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη και να δουλέψει με θεμέλιο με βάση τον κύκλο ζωής των υλικών. Και έτσι θα ενδυναμώσουμε την οικονομία μας και την πιο ανταγωνιστική. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά με τρόπο i4 και να τα ξαναβάλουμε στον κύκλο της οικονομίας με μια ολοκληρωμένη, σφαιρική προσέγγιση. Σχεδιασμός, παραγωγή, διανομή, κατανάλωση και επεξεργασία των αποβλήτων. Ακριβώς, όπως είπε ο Πρόεδρος, μια τέτοια φόρος ε, διαχείριση ήταν ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην ε, Γάνδη κατά αυτή την διήμερη άτυπη συνάντηση. Ο κύριος ε, Λάινεν παρέστησε αυτή την συνάντηση. Με την ευκαιρία θα πρέπει να το ξανά ευχαριστήσω για τη συμβολή του στην εκεί συζήτηση. Θεωρώ ότι το άτυπο αυτό συμβούλιο ήταν μια διοργάνωση πετυχημένη. Αυτές οι προσπάθειες για τη διαχείριση των υλικών είναι κάτι το οποίο γίνεται στα πλαίσια τις προσπάθειες για μια πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων στην Ευρώπη. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι υπάρχει ο χάρτης πορείας για το 2011. Το Δεκέμβριο το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει ότι θα γίνει στη συνέχεια επί τη βάση αυτού του χαρτιπορίας Επίσης, έχουμε και την ε, οδηγία που αφορά τα ε, απορρίμματα που προέρχονται από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη και συσκευές. Θέλουμε να υπάρξει πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο. Ήδη η Προεδρία έχει μελετήσει τις ε, τροπολογίες σας. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στην πρώτη αναγνώση. Θα ήθελα να σας πω δύο για την βιολογική επεξεργασία των ε, απορριμμάτων. Η προσέγγιση μας στην προσέγγιση βασίζεται στον κύκλο ζωής των υλικών. Έχει τονίσει η Προεδρία το ότι πρέπει να υπάρξει μια οδηγία για αυτό το θέμα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει προτάσεις σχετικώς. Τελευταίο στόχος, τελευταία μας πρόκληση είναι καλύτερα μέσα για την άσκηση της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος. Καλύτερη πραγματική της νομοθεσίας σημαίνει καλύτερη πολιτική το περιβάλλον. Καλύτερη προπαρασκευή, περισσότερες μελέτες επιπτώσεων και περισσότερα κίνητρα και καλύτερη χρήση αυτών των μέσων πολιτικής για το περιβάλλον. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η διακυβέρνηση του, της πολιτικής για το περιβάλλον για την διεθνή περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Επίσης, έχουμε ένα πρόγραμμα το 2012 που ενδιαφέρει και το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι θα βοηθήσετε την όλη προβληματική. Τώρα πέρα από τις ε, οδηγίες για τις ηλεκτρικές συσκευέ και τα επικίνδυνα υλικά έχουμε την νομοθεσία για το εξωτερικό του άνθρωπο σε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο που θα πρέπει να λάβει υπόψη τι έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι εξελίξεις έχει η δική σα εδώ προβληματική. Οπότε, κυρίε και κύριοι, για να μπορέσουμε για όλου αυτού του στόχου να σημειώσουμε κάποια πρόοδο, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σα. Γιατί ό,τι έχει πετύχει η Ευρώπη έχει βασιστεί στην συνεργασία και στο διάλογο. Έχουμε του επόμενου 6 μήνε πολλά να κάνουμε στον πρώτο περιβάλλον και ω Προεδρία Είμαστε έτοιμοι να ανταλλάξουμε τι απόψεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι νομίζουμε ότι θα είμαστε πιο συνεπείς στην πολιτική μας και ότι ε, θα έχουμε αίσια κατάληψη προστασία μας και ότι θα είναι αγαστή η συνεργασία μας μαζί σας. vielen Dank, Frau Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε για την παρουσίαση του προγραμματό σα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα και το γεγονό ότι προσπαθείτε να συνδυάσετε τις θέσεις του Συμβουλίου και του ε, Κοινοβουλίου προκειμένου να εξασφαλιστεί συμφωνία στα πιο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, τον κανονισμό για τα ηλεκτρονικά, τα ελαφρά οχήματα. Μακάρι. Η Υπουργοί από ό,τι ακούσαμε, ακούσαμε ναι, το Κανκούν, τη στρατηγική και τις τακτικές μπορεί να επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά αυτά θα εξαρτηθούν και από τα όσα πράττουμε εμείς. και την επιλογή για λόγους προστασίας των δικών μας συμφερόντων να ακολουθήσουμε μια οικονομία με χαμηλή, χα, χαμηλό άνθρακα. Ανεξαρτήτως τι κάνουν άλλοι. Και επίσης, ίσως θα ήταν σκόπιμο με τη συλλογή όλων των ηλεκτρονικών αυτών απορριμμάτων και άλλων ε, μηχανών, μηχανημάτων, να δούμε πόσο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα συλλέγουμε και να τα αξιοποιούμε. Θα ακούσουμε τώρα τους συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες, με πρώτα τον κύριο Ρίχερτ Ζέβορ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά βλέπω εδώ Περιφερειακή Υπουργό στην Προεδρία. Εγώ από το Τυρόλο που κατάγομαι και που έχουμε βέβαια πολύ έντονο τον ε, τοπικό χαρακτήρα και την ε, τοπικιστική νοοτροπία πρέπει με χαρά και εσάς εδώ ως Φλαμανδί Υπουργό. Αυτό που με εντυπωσιάζει κυρία Υπουργέ είναι ότι ξεκινώντας ε, την ομιλία σας και γνωστή Υπουργός Περιβάλλοντος μιλάτε για την οικονομική κρίση Λέτε δηλαδή κι εσείς ότι έχουν ε, στενό, στενή συνάφεια μεταξύ τους αυτά τα δύο φαινόμενα. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι είναι η καλή περιβαλλοντική πολιτική το κλειδί ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή αποδεικνύεται ούτως ή άλλως και ότι όλοι οι άλλοι πάνε στραβά και ότι οι δικές μας πολιτικές είναι ορθές, οι περιβαλλοντικές επιλογές. Τα κράτη τα οποία έχουν πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων τους είναι αυτά που έχουν και θα έχουν στο μέλλον ακόμη περισσότερο επιτυχία και ανταγωνιστικότητα. Επίσης, περιφέρειες. Για τις περιφέρειες το αναφέρατε και εσείς. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εφαρμογή σε παραδείγματι στην οδηγία για την προστασία των πτηνών ή για την προστασία της κλωρίδας και της πανίδας. Βλέπουμε πολύ διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές, περιφέρειες. Σκοπεύει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι φαίνεται ε, μάλλον σκοπεύει η Βελγική Προεδρία να πιέσει για να ενισχυθεί αυτή, αυτός ο βαθμός υλοποίησης της νομοθεσίας έτσι ώστε προς τα πάνω να προχωρήσουμε σε εξίσωση των ε, επιπέδων αυτών υλοποίησης και όχι προς τα κάτω φυσικά. Για το Κανκούν επίσης ε, γίνεται λόγος για μια χρηματοδότηση του τύπου fast track, ταχείου, ταχεία χρηματοδότηση, δηλαδή ταχεία τύπου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να διατηρηθούν και να τηρηθούν όπως πρέπει οι υποχρεώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά για τα ύδατα. Θα επισημάνω ότι περιμένουμε να δούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νέα οδηγία για το πόσιμο είδωρ, υπόσχεση την οποία έχουμε δει εδώ και ένα χρόνο, δυστυχώς δεν βλέπουμε να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει αυτές τις προτάσεις μας έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις Υποβάλλει πλέον. Πρόεδρος βεβαίως, ναι, τέτοιες ερωτήσεις για τα είδα τα πάντοτε ακούμε από εσά. Ευχαριστώ. Ο επόμενος συνάδελφος παρακαλώ όμως τηλεοράση να φύγει, δεν τους βλέπω κιόλα. είστε μπροστά μου. Παρακαλώ κυρία Μακάβνου. Ευχαριστώ την Υπουργό που ήρθε σήμερα και που μας μίλησε για τις ευαισθησίες της Προεδρίας της και για τα σημαντικά θέματα που τους απασχολούν για τους επόμενους μήνες. Μιλήσατε για το πρόγραμμα, το Κανκούν βεβαίω ξέρουμε ότι το έχουμε μπροστά μα. Μιλώντα με του Αμερικανού ότι μιλούμε χωρί πάντοτε να ε, προχωρούμε σε υλοποίηση, σε πράξη. Η Ευρώπη οτι μιλουμε χωρί παντοτε να προχωρουμε σε υλοποιηση σε πραξη η ευρωπη πίνη, υποστηριζει το στόχο του 30%. Διαρκώ αυτό λέει. Ε, όμως πριν από το Κανκούν μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα και ξέρω βεβαίω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το καθήκον της παρακολούθησης υλοποίησης και της διεκδίκησης μιας αποτελεσματικότερης εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Αλλά έχει τύχει ποτέ στο, Συμβούλιο Υπουργή των ε, ε, του περιβάλλοντος να ρωτούν ο ένας τον άλλον τι έγινε με αυτό το στόχο, με εκείνον το στόχο, τι έχει κάνει στη χώρα σου, τι σκοπεύεις να αλλάξει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις τα συντηρούν. Ε, ή μπράβο έκανες μια καλή, ανέλαβες μια καλή πρωτοβουλία πριν από δύο χρόνια κτλ. Ή στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είπε εκείνο, έκανες το άλλο. Γιατί είδαμε πόσο είχε αντισταθεί η αυτοκινητοβιομηχανία, ειδικά σε διάφορε προτάσει για πιο καθαρά αυτοκίνητα, και τώρα είναι εκείνοι που πρώτοι έρχονται να προβάλλουν νέα ε, ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ε, τι κάνει ο ένας και τι ο άλλος. Είναι καλό να ενημερωνόμαστε και να βλέπουμε βεβαίως και αν υλοποιούνται τα υπεσχημένα ή αλλιώς εάν απλώς λέμε λόγια του αέρα. Άλλη μια ερώτηση. Στα τρία, στους τρεις επόμενους μήνες η Επιτροπή θα κοιτάξει το θέμα των οροσίμων, το benchmarking δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτή τη στιγμή το απασχολεί μόνο τις Επιτροπές των Εθνικών Πραγματογνωμόνων. Πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι στο benchmark, αλλά αυτό φυσικά έχει και επιπτώσεις προς τις τιμές του άνθρακα. Το γνωρίζουν αυτά τα κράτη-μέλη και σε ποιο βαθμό. Όταν έρθει η ώρα να συζητήσετε το benchmarking. σε ευχαριστώ. Εκχαούτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν, μπορούμε, δεν έχω όρεξη να μιλάω κάθε μέρα Ολλανδικά. Σήμερα όμως θα υποφεληθώ και θα μιλήσω στα Ολλανδικά, επειδή υπουργό είναι και αυτή η Ολλανδόφωνη. Θα αναφερθώ σε δύο σημεία. Αναφέρετε τις τέσσερις προτεραιότητές σας αλλά για μένα όλα αυτά ακούγονται ακόμα πολύ γενικά. Θα ήθελα να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Δύο παρατηρήσεις λοιπόν. Πρώτον, μιλήσαμε για το κλίμα και το Κανκούν. Είπατε ότι θέλετε να έχετε μία θέση της Ένωσης. Καλώς. Λέτε όμως η Ένωση να μιλάει με μία φωνή. Το timing όμως δεν ήταν καλό. Η επιλογή του χρόνου δεν ήταν σωστή στην Κοπενχάγη. Δηλαδή, συμφωνήσαμε αρκετά πιο πριν, αλλά οι θέσεις είχαν αποφασιστεί από πριν, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Λέτε ότι θα έχουμε με τη θέση την Ευρωπαϊκή για το Κανκούν. Λέτε θα το βάλουμε στην ημέρη σε διάταξη. Εγώ τι λέω. Λέω ορισμένες από τις θέσεις μας, παραδείγματος χάρη μείωση κατά 30% των εκπομπών κλπ. Μην τα αφήνουμε για την τελευταία μέρα, την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου. Μιλήστε για την ε, αποσύζευξη, για τη Γάνδη, για την απόλυτη αποσύζευξη. Χρειαζόμαστε απόλυτη αποσύζευξη όσον αφορά τη χρήση των υλικών. Αυτό είναι ότι είμαστε πολύ στα γενικά, να περιμένουμε το 2011 ένα φύλλο πορεία εκ μέρου τη Κομισιόν. Όχι, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και άμεσα μάλιστα. Δηλαδή στην Ευρώπη να δώσουμε κίνητρα για την καύση των απορριμμάτων. Δεν κάνουμε την οδηγία για, για τα ανανεώσιμα. Χρειάζεται μια ιεράρχηση τι θα κάνουμε με τα απόβλητα και η αποτέφρωση είναι μια από τις τελευταίες βαθμίδες. Ζητάτε από την Κομισιόν ένα σχέδιο οδηγίας. Η Κομισιόν δεν θέλει όμως οδηγία για τα βιοαπόβλητα. Για την βιώσιμη διαχείριση των υλικών υπάρχει ένα τίμημα. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή μελετάει την οδηγία για την φορολόγηση της ενέργειας και εγώ θα σας ρωτήσω, θα ενθαρρύνετε την Κομισιόν σύντομα να μας παρουσιάσει αυτή την αναθεώρηση? Να μην πληρώνουμε με βάση την ποσότητα των όγκων, αλλά με βάση τη χρήση ενέργειας και τη ρήπανση. Να είστε λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένοι. Διαφορετικά θα περιμένουμε αυτό το φύλλο πορείας για πάρα πάρα πολύ καιρό θα είναι κρίμα για την Προεδρία σας. Πρόεδρος σας. Εγώ βέβαια θα έλεγα ο Ολλανδό βουλευτής να μιλάει Ολλανδικά ακόμα και αν δεν υπάρχει Φλαμανδός υπουργό μέσα στην αίθουσα. Καλό θα ήταν. Η κυρία Ρόσπαχ. Er Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. και με τον συνάδελφο μίλησε λίγο πριν από μένα και με τον σοσιαλδημοκράτη συνάδελφο. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Το να κάνουμε μία οδηγία μετά την άλλη χωρίς να ξέρουμε ποια θα είναι τα πρακτικά αποτελέσματα δεν είναι σωστή λύση. Όλο και περισσότερα χαρτιά και έγγραφε επί εγγράφων αυτό κάνουμε. όσον αφορά την αποτέφρωση των απορριμμάτων. Η... Τα μηχανήματα τρίτης γενιάς, όπως τα λέμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι πόρους δυνατούς διαθέτουμε, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και μιλάω για μικρά πράγματα, τα οποία όμως μπορούν να επιφέρουν αλλαγές. Να αποφεύγουμε αυτή τα τα βουνά ολόκληρα από πλαστικά σκουπίδια τα οποία ζούμε. Αυτά τα συζητήσαμε και με τον κύριο Επίτροπε. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα. Αντελβώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή που μας κάνει και το ότι ήρθετε. Η Ευρώπη θεωρεί το Ευρωκοινοβούλιο σαν ένα κινητήριο για τα θέματα του περιβάλλοντος, ίσως λίγο λιγότερο μετά την Κοπενχάγη. Ας ομολογήσουμε ότι ορισμένες χώρες μέλη δεν έδειξαν τη βούληση που χρειάστηκε να δείξουν όπως είχαν δείξει στο παρελθόν. Βέβαια, από τη μια μεριά δεν μπορούμε να αγνοούμε την δύσκολη οικονομική συγκυρία και να είμαστε ρεαλιστές. Από την άλλη μεριά όμως, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Σιμπέρ, δεν μπορούμε να αφήσουμε να μειωθούν οι φιλοδοξίες μας και να μην τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας και του Κανκούν και της Ναγκόγια. Η βιοπικιλότητα είναι μια τεράστια πρόκληση, το είπατε, και χαίρομαι που είναι στις προτεραιότητές σας. Είπατε επίσης ότι οι δεσμεύσεις που έχουμε λάβει είναι πολλές. το Γκέτενμπουργκ του 2001, τη διάσκεψη του Ιωχάνεσμπουργκ για τη Γη του 2002, το πρόγραμμα για τη βιοπικιλότητα 2006 και τις δεσμεύσεις του Μαρτίου φέτος του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, τα είπαν και οι συνάδελφοι, πώς η Βελγική Προεδρία θα μας διασφαλίσει ότι αυτή τη φορά η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα πραγματικά θα εφαρμοστεί. Τι συγκεκριμένες δεσμεύσεις, κατά τη γνώμη σας, και θα ήθελα να μας πείτε τη θέση σας, θα ληφθούν στη Βελγική Προεδρία και αυτές τις δεσμεύσεις θα τις ε, δώσετε γραπτά στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και επειδή η βελική αντιπροσωπεία θα είναι με την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην Αγκόγια, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το θέμα της δίκαιης πρόσβασης και στον επιμερισμό των πόρων, το περίπου πρωτόκολλο ΑΜΠΕΣ και ποιους, ποιοι είναι οι στόχοι σας σχετικά. Και μια τελευταία ερώτηση. Στην Επιτροπή μας τελευταία το έχουμε συζητήσει πολύ σχετικά με τις γενικά τροποποιημένους οργανισμούς. Φαντάστηκα ότι θα ασχοληθείτε με το κείμενο της Κομισιόν. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κατλίν Φαμπάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συνήθως μιλάω στη μετρική μου γλώσσα. αλλά του κάνουμε ιδιαίτερη ευχαρίστηση σήμερα. Θα επανέλθω στις δύο προτεραιότητές σας, από είπατε. Το ένα αφορά το κλίμα. Μία από τις προτεραιότητές σας είναι έκπληξη, αλλά ενδιαφέρον, είναι η βιώσιμη διαχείριση των υλικών. Θα αρχίσω με το κλίμα. Όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Πρώτον, οι στόχοι σας μιλήσετε για μια ε, προσωρινή προσφορά της Ένωσης όσον αφορά το 30%. Εγώ δεν συμφωνώ και υπάρχουν και άλλοι που δεν συμφωνούν. Εγώ θεωρώ μια Προεδρία θα πρέπει να αναζητήσει ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αυτό είναι το κύριο έργο σας βέβαια. Αλλά μια Προεδρία επίσης οφείλει να τολμά να κινείται προς μεγαλύτερες φιλοδοξίες όπως έκανε η Ισπανική Προεδρία. Ξέρουμε ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχουν 27 χώρες, το ξέρουμε και είναι... αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Πρέπει όμως να προωθούνται οι φιλοδοξίες μας και θέλω να ξέρω ποιες είναι οι δικές σας φιλοδοξίες. Δεύτερον, κάτι που επίσης είπατε, πρέπει να έχουμε αποτελέσματα και πρέπει να τολμούμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας. Μη σας παραξενεύει για μια συζήτηση που έγινε στην Κομισιόν. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο για το Περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει και άλλα συμβούλια. Ε, λοιπόν, πρόκειται για τη συζήτηση στην Κομισιόν του να δοθούν ε, επιχορηγήσεις για την εξόρυξη του άνθρακα. Αυτό είναι το ενεργειακό κοκτέιλ του μέλλοντος. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, το μέλλον δεν έχει θέση ο άνθρακας είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε ως εξόρυξη. Θα ήθελα λοιπόν το Συμβούλιο Περιβάλλοντος να είναι συγκεκριμένο στα μηνύματα που εκπέμπει. Να πει ότι για τις σπάνιες πρώτες ύλε στα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιούνται διαφορετικά. Γιατί μιλάμε για τρία δις, μιλάμε για τεράστιες επιδοτήσεις που δίνουν οι κυβερνήσεις και αυτοί τα τρία δις μπορούν να πάνε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οπότε θα πετυχαίναμε πιο γρήγορα το στόχο του 30% η βιώσιμη διαχείριση των υλικών συμφωνώ απόλυτα έχω γράψει ολόκληρα κεφάλαια για το θέμα αυτό είναι κάτι που ε, αφορά οπωσδήποτε το μέλλον και καλό είναι να το προωθήσει η Βελική Προεδρία όμως αυτό πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο στα επιμέρους, στους επιμέρους φακέλους. Έχετε οι συνάδελφοι Ρος και Φλωράνς αναφέρθηκαν στην οδηγία Φλωρέν, συγγνώμη Όχι εδώ είναι. Είχε πει ότι θα φύγει. Εμείς λοιπόν θέλουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Πιστεύω ότι γίνεται αυτό Στη Βελγική Προεδρία όμως πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση αυτή δεδομένου ότι με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει να υπάρξει άνοιγμα, δηλαδή στο θέμα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη βεντάλια ας το πούμε. Για την οδηγία ο Ιερός εγώ απογοητεύτηκα από τη θέση του Κοινοβουλίου να βγουν παραδείγματος τα ηλιακά κάτωπτρα από το πεδίο εφαρμογής. Καλό θα είναι το Συμβούλιο να πάρει θέση για τα ηλιακά κάτωπτρα που να είναι πιο ε, σύμφωνοι με την ε, βιώσιμη διαχείριση των υλικών. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και θα ακούσουμε βεβαίω τις απαντήσεις. Έτσι, θα έχουμε εξαντλήσει σχεδόν όλους τους, ερω... όλους τους ε, φλαμανδούς και Βέλγους με τον κύριο Στάση. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε για το θέμα των κλιματικών αλλαγών καταρχάς. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν λαμβάνεται θέση. Παραδείγματι τα βιοκαύσιμα όπου γνωρίζετε ότι πολλοί λόγος γίνεται, ότι είναι ένα ακαθόδες θέμα. Ότι μεγάλο μερίδιο της γης χρησιμοποιείται. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ε, βιωσιμότητας αυτού του συστήματος, γιατί το 1 τρίτο των εδαφών δεν λαμβάνονται υπόψη Και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε για, σε σχέση με την ε, βιωσιμότητα της βιομάζας ως συστήματος, αν είναι κάτι που θα θέσετε στο Συμβούλιο, εάν ε, η έμεση χρήση των εδαφών ή μάλλον απορρόφηση εδαφών για τη βιομάζα είναι κάτι που απασχολεί το Συμβούλιο, αν πρόκειται να το θέσετε. Γιατί εμείς το βλέπουμε ως πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό. Και νούμερα προβλήματα στο του, με το διοξείδιο του άνθρακα, εάν δεν λάβουμε υπόψη αυτή τη διάσταση, ε, είναι κάτι, όπως έλεγα, που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο για να δώσουμε τις απαντήσεις, λέει ο Πρόεδρος, εάν ε, είστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στις απαντήσεις για τον πρώτο γύρο τουλάχιστον των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί βουλευτές, για τα όσα είπατε και για το ενδιαφέρον το οποίο επιδείξατε για τις φιλοδοξίε μας, για τις ε, πρωτοβουλίες μας, για τις προτεραιότητές μας. Ε, οι προτάσεις σας και οι ιδέες σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ας ομαδοποιήσω τις ε, ερωτήσεις και ας αρχίσουμε με τα όσα είπατε σε σχέση με το κλίμα. Όντως η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις μεγάλες μας ε, προτεραιότητες και προκλήσεις. Ε, απέτυχε η Κοπενχάγη. Όμως θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Τελικά κάποια πράγματα εκεί συμφωνήθηκαν και με αφετηρία. Τα όσα συμφωνήθηκαν θα πρέπει να προχωρήσουμε και στους αντίστοιχους τομείς να σημειώσουμε πρόοδο. Ε, η βασική μας πρόκληση είναι το τι θα κάνουμε στην Κανκούν, όπου και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποια συμφωνία δεσμευτική και να δούμε τι θα συμφωνηθεί εκεί πέρα, το οποίο γενικότερα είναι δεσμευτικό γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εμείς θα είμαστε πρωτοπόροι, εμείς θα κρατάμε το πιδάλιο να προσέξουμε τη διαδικασία αυτή να προχωρήσει, να πιάσει τόπο, να μην αποτύχει. Βέβαια έχουμε βάλει τον πηγή ψηλά. Και από την άλλη μεριά, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, κατηγορούν εμά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ακριβώ συνέβη και στην Κοπενχάγη. ό,τι δεν πήγε καλά στην Κοπενχάγη με τις προσδοκίες, ε, για όλα έφταιγε, είπανε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την καταστροφή των δασών, ε, και τα άλλα θέματα τα, μας και θα πρέπει να τα εξετάσουμε, να δούμε τι γίνεται και με τον άνθρακα. Επίσης να δούμε την χρηματοδότηση γρήγορης εκκίνησης. Θα πρέπει και αυτό το θέμα το προωθήσουμε. έχουμε 2,4 δις ε, που προβλέπει να πάνε στο περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ECOFIN εξετάζει τη σχετική έκθεση. Θα πρέπει να δούμε με ποιου όρου και προποθέσει θα γίνει αυτή η ταχεία χρηματοδότηση. Όσο αφορά τώρα την πρόταση για τον περιορισμό των εκπομπών κατά 30% που έχει μπει σαν όρους και προϋπόθεση ανέφερα στην εισήγησή μου ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το να προχωρήσουμε προς τον στόχο αυτό των περισσότερων των εκπομπών εάν το κάνουν και άλλες χώρες και τα είπαμε στην ανακοίνωση. και ότι στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα συζητήσουμε αυτή την προϋπόθεση της περικοπής των εκπομπών. Τι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να πω ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο βρισκόνται στο ίδιο μήκο κύματο. Για την βιοπικιλότητα τώρα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Προετοιμάζουμε και πάνω σε αυτό το θέμα αυτό που θα ζητηθούν στο Θεοπορεινό Συμβούλιο. Να έχουμε κάποια θέση στο Μόντρεαλ ακόμα έχουμε κάποια πράγματα που συζητώνται και θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα προετοιμαστούμε. οι έχουν είπαμε, οι συζητήσεις για το Access and Benefit Sharing, το ABS. Η χρηματοδότηση βέβαια εδώ είναι το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα και επομένως το Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα και στο φθινοπορεινό συμβούλιο. Στη φθινοπορεινή σύνοδο. Επίσης, 15 Μαρτίου ελήφθη κάποια απόφαση, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε το πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις στο Μαντριόλ. βασικό ερώτημα είναι τι θα γίνει, ε, πώς θα εντάξουμε σε όλες τι πολιτικές την ε, μέρημνά μας για την βιοπικιλότητα, α πούμε στην ε, κοινή πολιτική και στην αλληλευτική πολιτική. Νομίζω ότι θα γίνει. Αυτό θα εξεταστεί και αυτό. Η κυρία Μάκαβαν μας μίλησε για το benchmarking. Συνήθω αυτά τα κανονίζουν οι επιτροπές, δεν πάει στο, πάνε στο Συμβούλιο. Το ίδιο αφορά ε, και στην ε, οδηγία για το νερό ε, όπου συζητήθηκε στην Τρόικα και έχουν γίνει κάποια βήματα πρόοδο για το πόσιμο νερό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε αφετηρία την σχετική οδηγία και να προχωρήσουμε από εκεί. Επίσης μιλήσαμε και για την ε, αηφόρο διαχείριση των υλικών. Έχουμε πάνω σε αυτό συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε το χάρτη πορείας. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για έγγραφα. Έχουν γίνει και συζητήσεις έχει συζητηθεί και το τι δράσεις συγκεκριμένες θα αναλάβουμε. Αυτά λοιπόν τα βρείτε και στο διαδίκτυο. Ε, τόσο και έχει αναφέρει η Προεδρία. Το ίδιο αφορά και για το οικολογικό σήμα, την, τον οικολογικό σχεδιασμό, όσον αφορά επίσης τη διαχείριση των ε, αποβλήτων. το ίχνος τον υγωγό του άνθρακα επίσης πρέπει να το ξανασυζητήσουμε την ανακύκλωση οπότε θα αναζητήσουμε κάποια λύση του τι μπορεί να γίνει για την πιστοποίηση σε σχέση με την ανακύκλωση μπορούμε βεβαίως να θέσουμε κάποιους στόχους και να εξεταστεί πώς μπορούμε ακόμα καλύτερα να εφαρμόσουμε τα όσα αποφασίζουμε. Η Σύνοδος του Δεκεμβρίου πρόκειται να δημοσιεύσει κάποια συμπεράσματα και ε, πάρα πολύ μας βοήθησαν τα όσα συζητήθηκαν στην Σύνοδο της Γάντης αυτό για τα βιοκαύσιμα, κύριε Στάση, ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Θα ζητηθεί το θέμα στην σύνοδο του Δεκεμβρίου. Πολύ σημαντικό για το περιβάλλον και θα πρέπει βέβαια στο Συμβούλιο να συζητηθεί και πάλι μια που έχουμε ένα σωρό θέματα που πρέπει να συζητηθούν και που κατατείνουν στην διαχείριση όπως τη θέλουν. Να είναι βιώσιμο. Στα αγγλικά. Εάν δεν απάντησε όλες τις ερωτήσεις, ξαναρωτήστε με. Κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις ακόμα βέβαια. Εν τω μεταξύ σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Okay. Ευχαριστώ πολύ και ε, ευχαριστώ... Ε, πολύ και ευχαριστώ την Υπουργό ε, Περιβάλλοντος που είναι εδώ παρούσα. Θα μιλήσω και εγώ τη μευρική μου γλώσσα, αυτή τη μειονοτική σχεδόν γλώσσα. Και θα ρωτήσω για τον προϋπολογισμό, αλλά με κάπως πιο ομούς όρους. Η Βελγική Προεδρία μας έχει πει ξεκάθαρα ότι πρόκειται να ασχοληθεί με το περιβάλλον περισσότερο κτλ. Και ακούμε διάφορα. Αλλά ό,τι και να κάνουμε χωρίς μέσα, μέσα διαθέσιμα δεν μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν ένας αγώνας, πρέπει να αποδεθούμε σε έναν αγώνα για το περιβάλλον και στην ε, περιβαλλοντική μεταρρύθμιση που δεν προσφέρεται κάθε δεν προσφέρεται πάντοτε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς ε, η Βελγική Προεδρία σκοπεύει να συζητήσει τα θέματα του προϋπολογισμού, τα δημοσιονομικά, με τρόπο ώστε να γνωρίζουμε όλοι το τι κάνουμε να μπορούμε να ε, χρηματοδοτούμε και το Life Plus και άλλα τέτοια προγράμματα ε, με επαρκή κονδύλια. Διαφορετικά δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερνάνδες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, με συγχωρείτε πρόεδρε που άρχισα να λάβω το λόγο, αλλά ακούω ακόμα τη ερμηνεία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί το πρόγραμμά σας είναι φιλόδοξο. Μιλήσατε για αποτελεσματικότητα, για βιώσιμη ανάπτυξη και μιλήσατε και για συγκεκριμένες δράσεις. Φαντάζομαι η, κρίση που, η οικονομική κρίση που ζούμε θα είναι ένας κίνητρο να κινηθούμε προς μια κοινωνία περισσότερης ανακύκλωσης με έννοιες απόδοσης που θα πρέπει να ορίζονται και ως προς το περιβάλλον. Υπήρξε εισηγητής για τα βιοαπορρίμματα. Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο. Και χαίρομαι για το ότι είπατε ότι ελπίζετε η Κομισιόν να κάνει πρόταση οδηγίας Εγώ από τη Βελγική Προεδρία περιμένω μια συγκεκριμένη φιλοδοξία στο θέμα αυτό. Μην περιμένουμε η Κομισιόν να μας παρουσιάσει ένα έγγραφο. Πρέπει να ασκήσετε πίεση. Η Κομισιόν μιλάει και λέει αντιφατικά πράγματα στο θέμα αυτό. Από τη μια μεριά θέλει μια νομοθεσία χωρί κενά και από την άλλη μεριά ο Επίτροπο μα λέει ότι χρειάζονται περισσότερε προδιαγραφέ. Παραδείγματο χάρη προκειμένου να έχουμε εναρμόνιση για αυτό που λέμε compost. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής. Και μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας για να προστευτεί το ε, σημερινό πλαίσιο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια διάσπαρτη νομοθεσία, διάσπαρτα κομμάτια ε, νομοθεσία σε διάφορα τμήματα και εμείς αυτό που θέλουμε είναι σαφήνια, βεβαιότητα, νομική βεβαιότητα που θα το είχαμε αν είχαμε μία μόνο οδηγία. Έπειτα, να είμαστε και φιλόδοξοι αλλά να είμαστε και ρεαλιστές. Γι' αυτό το να λέμε υποχρεωτική συλλογή των απορριμμάτων όπου είναι δυνατόν ναι αλλά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής οικονομική και περιβαλλοντική και σας ερωτώ τι συγκεκριμένο μέτρο έχετε κατά νου και ποια είναι η στρατηγική σας. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τη στρατηγική σας. Γιατί μερικές φορές το μυστικό είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε ή όχι αυτό που έχετε κατά νου πώς σκοπεύετε να προχωρήσουμε έτσι ώστε η κοινωνία αυτή ανακύκλωση που έχει πλέον εκτίματα όσον αφορά την καταπολέμηση στην αλλαγή του κλίματος για τη βιοποικιλότητα Η κομπόστ καλής ποιότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ποιότητα του εδάφους και για την καταπολέμηση της υποβάθμισης των εδαφών. Διαφορετικά θα έχουμε επιπλέον κόστος 30 και δις ευρώ Επιβάλλεται λοιπόν και για οικονομικούς λόγους να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να έχουμε μια οδηγία. Και επαναλαμβάνω, μπορείτε να υποστηρίζετε και στη δική μου πλήρη συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και Πρόεδρε του Συμβουλίου. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι συνδυάζεται δύο αρμοδιότητες οι οποίες συνήθως ε, δεν συντρέχουν πολιτισμός και περιβάλλον. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ούτω ώστε να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια, να κάνουμε την αλλαγή, δηλαδή για να μην έχουν τις εξαγγελίες ε, που είναι μεγάλα λόγια και ποτέ δεν είναι πραγματικότητα. Αυτό επίσης με χαροποιεί γιατί με ενδιαφέρει και εμένα και ο πολιτισμός και, και το περιβάλλον. Και απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίω ε, η υπόθεση των, της βιώσιμης διαχείρισης των υλικών. Πρόκειται επομένω τώρα για ε, ένα στόχο ε, πάρα πολύ καυτό θέμα και κυρίως όσον αφορά τον το, το, το κλάδο των ε, οικοδομών, τον κατασκευαστικό. Ε, χρειαζόμαστε να κάνουμε οικονομία όσον αφορά τα υλικά. Υπάρχουν κάποια στατιστικά τα οποία μας δείχνουν ότι πάμε για καταστροφή στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε ε, τα κατάλοιπα, έχουμε τα απορρίμματα, όλα, όλα αυτά τα οποία όταν γκρεμίζεται ένα κτίριο ε, δημιουργούνται και ε, έχουμε την ε, προφή, τη συντήρηση της αρχιτεκτονικής της παραδοσιακής αλλά επομένως έχουμε για τις ανοιχτέ πληγές που είναι ακριβώς όλα αυτά τα απορρίμματα και τα υλικά. Είναι το πιο σωστό να υπάρξει μια πρωτοβουλία για την αυτό αυτού του προβλήματος, κάτι το οποίο θα το αναδειχθούν και οι επόμενες προεδρίες. Υπάρχουν ένα σωρό μελέτες με πάρα πολλά στοιχεία το Princeton, το Πανεπιστήμιο έχει κατεβάσει μια τέτοια μελέτη με κάποιες προτάσεις και σε ΗΠΑ πολιτείες έχουν μια σωστή πολιτική ότι έχουμε 25% ε, περισσότερη απασχόληση από το κατασκευαστικό τομέα ε, με την αντιμετώπιση αυτήν σε σχέση με τη δική μας. Οπότε Έχουμε το πετρέλαιο και τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Αλλά όσον αφορά λοιπόν αυτή την προστασία των παραδοσιακών μνημείων πρέπει να το κάνουμε εμείς και όχι να έρθουν οι Κινέζοι να το κάνουν. Στο κάνουν κάποιες επιχειρήσεις τοπικές. Παρακαλώ η Προεδρία σας ας μπορέσει να κάνει μια τέτοια προσπάθεια νομίζω είναι πολύ σημαντικό, θα το στηρίξουμε εμείς και αυτό μπορεί να το συνεχίσουμε από όμως προεδρίες. Ευχαριστώ. Είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερο στην ε, συνάδελφο περιβάλλον και πολιτισμός, ιστορικά κτίρια και περιβάλλον. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα μιλήσω φλαμαδικά. Ευχαριστώ την κυρία Υπουργό. Είναι σημαντικό το ότι ήρθε. Κατά τη γνώμη μου, οι διαπραγματεύσεις έχουν κάπως βαλτώσει, διότι δεν δώσαμε πολιτική απάντηση, πολιτική πρόταση στη διακήρυξη του Μπαλίου, του Common Response ε, Differentiate but differentiated responsibility. Και ενώ δεν δίνουμε μια τέτοια απάντηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ομοφωνία, πράγμα το οποίο θέλουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και για την αύξηση της θερμοκρασίας και για τις ε, φυσικούς πόρους και πρέπει να ξέρουμε πρώτον ότι η φυσική πόρη είναι πεπερασμένη δεύτερον η ικανότητα της γης να μεταβολίζει τα απορρίμματά μας και αυτή είναι πεπερασμένη. Η αύξηση θερμοκρασίας έχει σχέση με την καύση των ε, ορυκτών καυσίμων που και αυτά είναι πεπερασμένα. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα σωστής διαχείρισης των υλικών. Πρέπει να πάμε πολύ περισσότερο στη ρίζα του προβλήματος. Δηλαδή, η φυσική πόρη είναι πεπερασμένη και πρέπει το πρόβλημα αυτό των φυσικών πόρων να το δούμε πολιτικά. Δεν ε, τεχνολογικό θέμα, πώς θα γίνει η καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών, αλλά να καταλάβουμε ότι αν είμαστε σοφοί στο να βρούμε ένα σύστημα διεθνούς διακυβέρνησης που να μας εξασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και για μας και για τις μελλοντικέ γενιές, θα καταλήξουμε σε κατάσταση σπάνης και εκεί ο πιο ισχυρός χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες που σημαίνει σειράξει. Για να είμαστε σοβαροί στη δράση μας. Ξαναγυρίζω στο θέμα της ε, αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να περάσουμε από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Πρέπει να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το πέρασμα. Δεν έχει νόημα να λέμε μείωση 20-30% όταν κάτι που έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν και πρέπει να το κάνουμε διότι αν καταφέρουμε να το κάνουμε με ένα αποτελεσματικό crash program θα έχουμε λύση και για την οικονομική κρίση που βιώνουμε. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ευθέως με πολιτικό τρόπο. Και εγώ είμαι στη διάθεση της Προεδρίας αν χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση. Πρώτος ευχαριστούμε. Η Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο, Προεδρεύουσα. Είναι ευρύ το φάσμα των τομάτων που μας παρουσίασε Χαίρομαι για την πολιτική συμφωνία που σκοπεύετε να προωθήσετε για τα βιοκτώνα και ρωτάω βεβαίως σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει το Συμβούλιο σε αυτή τη συμφωνία. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ή τουλάχιστον στην Επιτροπή μας έχουμε μια σαφή γραμμή. Πρόκειται να ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο, ε, αλλά είναι σαφές ήδη το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, μάλλον η τάση ότι θέλουμε σαφή κριτήρια, αυστηρούς κανόνες. Και όπου υπάρχουν εξαιρέσει να εφαρμόζονται με αυστηρότητα και να είναι σαφώς προσορισμένες. Ιδιαίτερα μας ε, απασχολεί η αηφορία, ε, η βιωσιμότητα, η προστασία των ε, ζώων, της ευημερίας των ζώων, γιατί δεν θέλουμε βεβαίως να εφαρμόζονται αυτές οι σειρές από πειράματα που προβλέπονται και στην οδηγία για τα βιοκτώνα πάνω σε ζώα. Θα θέλαμε λοιπόν να προσδιοριστούν με συγκεκριμένους όρους ποια είναι τα πείραματα που είναι άκρος απαραίτητα, ποια είναι εκείνα τα οποία περιτεύουν, μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε από κάποια άλλη λύση έτσι ώστε να έχουμε το ελάχιστο δυνατό σε πειράματα σε ζώα. Ο κύριος Ζέμπαρς μίλησε για τα πόσιμα ύδατα και, τη σχετική, και σχετικό κανονισμό. Ξέρω ότι υπάρχουν κράτη-βέλη τα οποία ανησυχούν διότι η ε, πρόταση για τα βιοκτώνα οδηγεί σε λύσεις ευρωπαϊκές, δηλαδή θα μπορεί το κάθε κράτος χωριστά να δίνει τις άδειέ του, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει η οργάνωση και θα πρέπει να δούμε και σε σχέση με, το, με την προστασία των υδάτων και τα πόσιμα ύδατα, τους σχετικές ε, διατάξεις και κανονισμούς, ε, πώς μπορούμε να έχουμε την, τον προσδορισμό των μεγάλων, των κύριων στόχων που θα ισχύουν για όλους. Και επίσης, ε, κυρία Υπουργέ, ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει όταν μιλούμε για μία ενιαία αδειοδότηση και έλεγχος του κόστους που θα συνεπιφέρει ε, η εφαρμογή της, γιατί ε, δεν μιλούμε στην περίπτωση των βιοκτώνων για μεγάλες επιχειρήσεις με ευρύ περιθώριο οικονομικό, αλλά για μικρές και μέσες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επιβαρυνθούν υπερβολικό κόστος. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Μπέλετ, για να τελειώνουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Υπουργό και σας εύχομαι καλή τύχη, καλή επιτυχία για όλες τις φιλοδοξίες και τις προτεραιότητες σε σχέση με την ε, μείωση των εκπομπών ε, και από τις μεταφορές και από τα ελαφρά οχήματα, ε, ελαφρά επαγγελματικά εμπορικά οχήματα. Πάντως αυτά τα οποία εκτέθηκαν δεν είναι αρκετά Βεβαίως και είναι σημαντική η μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές. Μακάρι να καταλήξετε σε κάποια συμφωνία στην Κανκούν. Όμως, αυτό είναι θέμα ενεργειακό, ε, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό για το περιβάλλον. Να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, υπάρχουν ε, ε, ιδέες για ε, να γενικευθεί η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών οχημάτων. Το ξεκίνησε, το συνέχισε τέλο πάντων και η Ισπανική Προεδρία. παρακαλώ εσείς, αν μπορείτε, επιβεβαιώστε ότι συνεχίζετε τις προσπάθειες και την πίεση να προχωρήσει η υπόθεση αυτή των ηλεκτρικών οχημάτων. Κάτι να υπάρχει του χρόνου, να είμαστε έτσι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για τις, ερωτήσεις, για τις ερωτήσεις. Πριν να περάσουμε στι απαντήσεις, θα να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Αμπράμι και τον καθηγητή κύριο Αμπράμι και όλη την ομάδα από τη Βενετία που θα ε, μας μιλήσουν ε, για το θέμα ενός ποινικού δικαστηρίου για περιβαλλοντικά εγκλήματα. Αλλά παρακαλώ τώρα την κυρία Υπουργό να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τις θετικές σας αντιδράσεις, για τις προτεραιότητες μας. Μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά σημαντικά θέματα υπόθηκαν. Όκερ, κύριε Όκερ, για τη χρηματοδότηση έχετε δίκαιο. Είναι βάσιμα τα επιχειρηματά σας. Περιβαλλοντική πολιτική σημαίνει και μέσα χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό, και το είπα νομίζω και στην παρουσίαση μου νωρίτερα, ότι πρέπει να προσδιορίσουμε καλύτερα την αξία. Αυτό που ονομάζουμε TEEB, ε, οικονομική δηλαδή αξία των οικοσυστημάτων μας. Γιατί αν μπορούσαμε να τα προβάλλουμε, ήδη θα είχαμε προχωρήσει σημαντικά. Και αυτό αποτελεί και για τον κύριο Ζήμπαχ μια, μια απάντηση που ε, έκανε την παρατήρηση ότι ξεκινώ με την οικονομική πολιτική για να φτάσω στην περιβαλλοντική. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε ξεκομμένα αυτά. Είναι ευκαιρία η οικονομική κρίση για να περάσουμε σε μια ε, οικονομία με χαμηλό άνθρακα. Και δεν πρέπει να περιμένουμε να περάσουν χρόνια για να το κάνουμε αυτό. Πρέπει αμέσω τώρα να το πράξουμε. Κάποιοι μιλούν για διέξοδο και για δημοσιονομικέ κρίσει. Ναι, αλλά η λύση θα είναι, πιστεύω, κράτατα η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Και αυτό ασφαλώ θα μα απασχολήσει στο Συμβούλιο. Για τα δύο απόβλητα. Με χαρά βλέπω ότι υπάρχει πρόταση του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσουμε να την προωθήσουμε. Γιατί ε, ο κύριο Κουτιέρης που μίλησε για την ε, διαχείριση των υλικών και την ε, διασύνδεση, το, το, τη συνάφεια με το υλικό. Ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να φτάσουμε στην ανακύκληση του ε, οικοδομικού υλικού, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε την ιδέα αυτή γενικά στην οικονομία μας. Όταν παρασκευάζουμε ένα προϊόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι ανακυκλώνεται. Και για τον κύριο Πρόντι, ο οποίο είπε ότι έχουμε περιορισμένο υλικό στη διάθεσή μας, πεπερασμένους πόρους και πρέπει να τους χρησιμοποιούμε οικονομικά. Θα το συζητήσουμε. Σημειώνα τόσο είπε η κυρία Κλάς για τα βιοκτώνα και την πολιτική συμφωνία σε επίπεδο συμβουλίου. Οδηγία για τα πόσιμα είδα την κάλυψα νομίζω. Και αν μου επιτρέπετε θα επανέλθω σε μια ερώτηση της κυρίας Εκχάουντ για το κλίμα, την, ε, τον έθετο χρόνο και την έγκαιρη στρατηγική που αναφέρατε. Ναι, ακριβώς γι' αυτό στο άτυπο συμβούλιο συζητήσαμε με την ε, βιώσιμη διαχείριση των υλικών, αλλά είχαμε και ένα γεύμα εργασίας για να συστήσουμε μια στρατηγική για το Κανκούν, ώστε να μην ε, πάμε απροετοίμαστοι. Είπαμε λοιπόν ότι συμφωνούμε να έχουμε κοινά μηνύματα, να είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, να λέμε το ίδιο πράγμα και είπαμε ότι θα οργανωθούμε με τις, μεταξύ μας οι αντιπροσωπείες ώστε να συνεννοούμαστε, να συναντιόμαστε και να ε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες ώστε να έχουμε μια κοινή παρουσία αυτά θα τα ξαναδούμε και θα τα υποβάλουμε στο, Γενικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Οκτώβριο, ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Αυτό είναι ο στόχο μα, εν πάση περιπτώσει, ο στόχο τη βελική Προεδρία. Και μια ερώτηση του κυρίου Μπελέτ, η τελευταία ερώτηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όπου πάλι έχουμε να κάνουμε την ανακύκλωση, με την αναδιάρθρωση της οικονομίας μας. Με, έχουμε να κάνουμε με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι καλύτερο και για τον τρόπο ζωής μας και για το περιβάλλον. Είναι πιο οικονομικό. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε και θα επιμείνουμε για να πείσουμε τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε, οι παρατηρήσεις και οι ερωτήσεις σας στους στόχους της Προεδρίας. Επανέρχομαι με την προσφορά μου να διατηρήσουμε επαφή και να συζητούμε όποτε χρειαστεί κάποιο θέμα. Είναι σημαντικό τα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη στις εργασίες μας στους επόμενους μήνες είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην τα συζητήσουμε, γιατί από κοινού πιστεύω θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, βλέπουμε με χαρά την στράτευση στον αγώνα αυτό για το περιβάλλον. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρετε στο εξάμεινο αυτό. Στην Αγκόγια και το Κανκούν το Κοινοβούλιο θα είναι παρόν με αντιπροσωπεία και έχουμε βέβαια μια πάγια, ένα πάγιο αίτημα που σε έναν βαθμό προκύπτει και από το, τη συνθήκη της Λισαβόνας να μας επιτραπεί η συμμετοχή σε, μάλλον να αναλάβουμε και εμείς το ρόλο μας και να συμμετάσχουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η αντιπροσωπεία πρέπει να παρτίσει όχι από Συμβούλιο και Επιτροπή, αλλά από Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Και τουλάχιστον οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών πρέπει να είναι παρόντες. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε πιστεύω. Συγχαρητήρια. Θερμά. Προς το παρόν. Και περνώ στο επόμενο θέμα. Μόλις χαιρέτησα τον καθηγητή κύριο Αμπράμι με την αντιπροσωπεία του που θα μας ενημερώσει για το θέμα, για την ιδέα ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα ο Δ. Φρένι Κρούναρτ καθηγητής Κόντι και ο Ρομπέρτο Αντώνη είναι παρόντες. Μια ιδέα που πηγάζει από τη Βενετία. Διεθνής Ακαδημία των Περιβαλλοντικών Επιστημών. Ιδιαίτερος χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ σήμερα. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Να μην χάσουμε καθόλου χρόνο λοιπόν και σας δώσω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Φερνάντες, ήδη έχουμε περάσει το επόμενο θέμα της ημερησής διάταξης. Αν έχετε κάτι να ε, εξαντλήσετε με τον συνάδελφό σα. παρακαλώ. Μπορείτε, εάν θέλετε, να έρθετε εδώ. Πολύ ευχαριστώ. Καλύτερα θα σας βλέπουμε κιόλας. Here. So, okay. So we start in Okay. So I give you the floor to present uh, yes, concise. Σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε στο δυνατόν πιο συγκεκριμένα τις προτάσεις σας. Ο κύριος Γκρούναρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας εδώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Επιτροπής Περιβάλλοντος, κύριο Γιολάινεν και όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν τα θέματα της ε, ε, ελευθερίας, της εγγύησης ελευθερίας ζωής για όλους μας ε, να μην υποβληθούν σε έναν αυτοκρατορικού τύπου ρελατιβισμό και να μην ε, συζητηθούν σε μια βάση τάμπουλα ράζα ε, επιστημοτεχνολογική, αλλά να προχωρήσουμε σε περαιτέρω προσπάθειες. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη κοινωνία εάν εγγυηθούμε το δικαίωμα σε ελευθερία, θεμητό δικαίωμα ελευθερίας βέβαια για τον κάθε έναν, αλλά ταυτόχρονα διαφυλάσσοντας και τον ε, πλούτο που εξασφαλίστηκε τους τελευταίους αιώνες μέσα από μια συλλογική ευθύνη για τον κάθε ένα, ευθύνη του ανθρώπου ενάντια της βιοσφαίρας. Και έτσι η Ακαδημία των Επιστημών του Περιβάλλοντος θέλει να, να προσφέρει στη διάθεσή σας ε, τις εμπειρίες της, τις γνώσεις σας με την ελπίδα ότι θα καταλήξουμε σε μία συνένεση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί τους οποίους περιμένουμε, δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο πια, εμείς πρέπει να λάβουμε δράση και δεν χρειάζεται να περιμένουμε πια. Αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, καταρχήν ευχαριστώ τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος, διότι μας ε, έκανε την τιμή. Να μας προσκαλέσει να αναφέρουμε για τα προγράμματά μας στην Επιτροπή σας. Επίσης ευχαριστώ τους ε, βουλευτές μέγη της Επιτροπής για την προσοχή που επέδειξαν και προς εμάς και προς τα προγράμματά μας. Μετά από την επιστολή 13 Μαΐου που έστειλε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και ως συνέχεια, κύριε Πρόεδρε Λάινεν, απευθύνεται άμεση πρόσκληση, έγιναν τα εξή. Πρώτον, γιατί χρειάζονται να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Τα προβλήματα λόγω της μείωσης των πώς επηρεάζουν οι πρώτες ύλες στην υγεία του ανθρώπου κλπ. Είναι κάτι γνωστό από πολύ παλιά. Αλλά η σχέση αυτή είναι μια σχέση μιας αμοιβαίας επιθετικότητας. Όπου δυστυχώς η επιθετικότητα μερικές φορές ε, από τη μεριά του ανθρώπου χαρτίζεται από δόλο. Και η τελευταία καταστροφή, φυσική καταστροφή με την έκρηξη στο πλατφόρμα offshore στις Ηνωμένες Πολιτείες μια ακόμα απόδειξη της σοβαρότητας του προβλήματος περιβάλλον και ότι επήγει η παρέμβασή μας κυρίως με ένα σύστημα ελέγχων και κυρώσεων που θα εγγυάται μια αποτελεσματική δικαιοσύνη. Έτσι στη συνείδηση των λαών υπάρχουν ήδη δύο δεδομένα τελείως αποδεκτά. Πρώτον, η ανάγκη να υπάρχει μια συντονισμένη νομοθεσία που θα βάλει αυστηρά όρια στις, στην ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπεριέχει δυνητικά μεγάλο κίνδυνο για το οικοσύστημα και υπερεθνικά όργανα καταστολής συμπεριφορών που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε περιβαλλοντικά εγκλήματα. Χρειαζόμαστε μια πιο, ε, πιο αποτελεσματικός έλεγχος των ρηπαντών και καλή χρήση των πρώτων υλών. Ορισμένα προϊόντα που θεωρούνται ασφαλή όπως ορισμένα φυτοφάρμακα κλπ. Τελικά είδαμε σε τι ανθρώπινες τραγωδίες οδηγήσαμε στον Ποπάλ με 500.000 θύματα και χιλιάδες χιλιάδες νεκρούς. Εξάλλου εδώ και χρόνια η, η επιστήμη έχει συνειδητοποιήσει αυτή τη σοβαρή κατάσταση και μελετάει με όλο και μεγαλύτερη προσοχή τα θέματα που αφορούν την υγεία του πλανήτη. Και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μας δείχνουν ότι πρέπει να βρεθούν κατάλληλες απαντήσεις στο πρόβλημα περιβάλλον. Μεταξύ των μελετών ας αναφέρουμε μία που έγινε με βάση της παρατηρήσεις από δορυφόρους χρήση δηλαδή ε, δορυφόρων της NASA και μετά αξιολογήθηκε στο, αναλύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το Φεβράριο του 2001 από 3.000 επιστήμονες επί τόπου για μελέτη του περιβάλλοντος του πλανήτη και να προτείνουν και λύσεις. Η ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκε ένας είδος χάρτης των καταστροφών του περιβάλλοντος. Ένας άθλαντας που βγήκε από μια παρακολούθηση που μας δείχνει μια πολύ ανησυχητική αλήθεια. Ο άνθρωπος μεταξύ του 1600 και του 2000 δημιούργησε καταστροφές για το περιβάλλον που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του πλανήτη Γη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που τη λέμε και την ξαναλέμε εδώ και χρόνια, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μια αρχή που ε, είναι καθολικής αξίας, γιατί έχει μπει στη συλλογική συνείδηση εδώ και καιρό και σε νομοθετικά κείμενα εδώ και 30 χρόνια. Αν δούμε τα τελευταία 30 χρόνια, βλέπουμε ότι πρωτεύουσες σημασίας είναι η περίοδος 72-92 όπου ορίμασε σιγά σιγά η συλλογική συνείδηση για τη σοβαρότητα του προβλήματος περιβάλλον που δεν θεωρείται πια ένα τοπικό πρόβλημα ή περιφερειακό ή και εθνικό καν είναι πρόβλημα πλανητικών διαστάσεων. Έπειτα έχουμε και αύξηση των επιστημονικών γνώσεων, νομικών και επιστημονικών γνώσεων και συνειδητοποίηση της ανάγκης να υπάρχει πρόληψη και καταστολή μια δικαιοσύνη που θα επιβάλλει κυρώσεις αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Και πρέπει να υπάρχουν ορισμένε βασικές αρχές γι' αυτό, προκειμένου να έχουμε τις μεταρρυθμίσεις και νέα υπερεθνικά εργαλεία. Η αρχή του οριπένων πληρώνει, να μην είναι σε βάρος δηλαδή της, του κοινωνικού συνόλου, η αρχή της πρόληψης, της βιωσιμότητας, της διόρθωσης της άρσης της αιτίας της ρήπανσης. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, για τους κύριοι βουλευτές, πρέπει να υπάρξουν προδιαγραφές για μια αποτελεσματική δικαιοσύνη με κυρώσεις, όπως είπα, αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τις κυρώσεις, να εφαρμόσουν ποινικέ κυρώσεις για εγκληματικές ενέργειες που είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και ο Εθνικός Δικαστής άμεσα πρέπει να κάνει αποτελεσματική έρευνα και ανάκριση ιδιαίτερα που υπάρχει δόλος στην καταστροφή ε, πυρκαγιές δασών στην Ελλάδα εμπρισμοί δασών άμεσα πρέπει να γίνει η ανάκριση για να αποδοθούν ευθύνες και μετά πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, ποινές. Υπάρχει ένα σχετικό ψήφισμα 14 Σεπτεμβρίου 2009. Επίσης, πρέπει να υπάρξει και ένα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το Περιβάλλον. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο για το Περιβάλλον. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις και γιατί προτείνουμε αυτό το ε, ποινικό δικαστήριο και τι πλεονεκτήματα θα έχει μια τέτοια κίνηση. Η μεταρρύθμιση θα μας επιτρέψει να πετύχουμε ταυτόχρονα πολλούς στόχους. Πρώτον, να ξανατογιστούν οι αρχές της αποτελεσματικής δικαιοσύνης, effective justice. Θα υπάρξει ένα νέο κοινωτικό όργανο που θα εγγυάται τον δικαστικό έλεγχο για τη χρήση και κατάχρηση των πόρων του περιβάλλοντος, μια ευρωπαϊκή ποινική δικαιοσύνη για το περιβάλλον πιο ομοιόμορφη σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση ήταν μια συμβολή από εμπειρίες και ιδέες και για τους λαούς της Μεσογείου, την ευρωμεσογειακή περιοχή δηλαδή, η Ένωση θα έχει βάλει το περιβάλλον στο κέντρο των ενδιαφερόντων της. Επίσης, η μεταρρύθμιση σε συμφωνεί με ένα αίτημα δικαιοσύνης εκατομμυρίων πολιτών της Ένωσης κάθε φορά που έχουμε μια κατάσταση ρήπανσης που συχνά μένει ατιμόρυτη. Στην περίπτωση Άουρουλ που κατέστρεψε το Δούναβι και η Ένωση διαπίστωσε ότι η τελευταία αυτή η ρήπανση του Δούναβι επιβεβαίωνε την ανυπαρξία συστήματος προστασίας των οικοσυστημάτων. 100.000 κυβικά μέτρα τοξικές λάσπη από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία κλπ. Τα ξέρουμε αυτά. Τρομερή τραγωδία οικολογική. Άλλος στόχος. Να αποφύγουμε καταστροφές στη θάλασσα. Πρεστής, έρικα, τεράστια ζημιά Και η ζημιά όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και στη βιομηχανία. Πάμε χάρη οι αλίες, ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία. Δεν είναι μόνο η ζημιά στην ίδια τη θάλασσα, τεράστια ζημιά για θέσεις εργασίας, για την ίδια την οικονομία πλήγμα. Οι μεταρρυθμίσεις επίσης θα οδηγούσαν σε παράλληλη κίνηση με την άλλη μεταρρύθμιση της Ένωσης με την Οδηγία 2008-99 του Συμβουλίου για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικών διαδικασιών. Και θα είναι υποχρεμένες οι χώρες μέλη να επιβάλλουν ποινικέ κυρώσεις σε εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος αυτό το επίπεδο εναρμόνισης θα επιτρέψει την εφαρμογή πιο αποτελεσματικά του δικαίου περιβάλλοντος με προστασία του περιβάλλοντος όπως προβλέπει εξάλλου το άρθρο 174 της Συνθήκης. Σας είπα όλα αυτά περνάνε ετοιμόρυτα μέχρι τώρα. Η Ένωση γνωρίζει και ότι όλοι και πιο πολλά τέτοιου είδους εγκλήματα υπάρχουν και όλο και περισσότερες απειλές. Και οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα κυρώσεων σε όλες τις χώρες. Η οδηγία που σας ανάφερα πριν για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου θα εγγυάται μια ομοιόμορφη ποινική προστασία υπέρ του περιβάλλοντος σε όλη την Ένωση. Όλοι ξέρουμε ότι η οδηγία εξασφαλεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας Το γεγονός ότι τα εγκλήματα αυτά αποτελούν απειλή για το περιβάλλον απαιτεί άμεση αντίδραση και η εμπειρία επαναλαμβάνω μας έχει δείξει και αυτό είναι σημαντικό και το τονίζω ότι τα συστήματα κυρώσεων που υπάρχουν, όχι οι ίδιες οι κυρώσεις, τα συστήματα των κυρώσεων που υπάρχουν δεν επαρκούν για πλήρη τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η τήρηση πρέπει να ενισχυθεί μέσω ποινικών κυρώσεων όπου η κοινωνία θα αποδοκιμάζει με τρόπο διαφορετικό από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα με διοικητικές και άλλου είδους τέτοιες κυρώσεις. Μια αποτελεσματική προσία του περιβάλλοντος απαιτεί κυρώσεις αποτρεπτικές για δραστηριότητες σε βάρος του περιβάλλοντος γιατί όπως ξέρουμε όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα μέχρι τη στρατόσφαιρα, της γης, της χλωρίδας, της πανίδας και τη διατήρηση των ειδών. Παράλληλα με αυτή την υπόθεση μεταρρύθμισης που σας ανάλυσα και μπορούμε να συζητήσουμε, υπάρχει μια άλλη υπόθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Περιβάλλον. Αυτό είναι πιο πολύπλοκο θέμα ως πρόταση ως υπόθεση. Αλλά η, η, Ακαδημία μας προωθεί την ιδέα αυτό εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Και η επικαιρότητα της οδηγίας τονίζει την υποχρέωση των κρατών να επιβάλλουν κυρώσεις σε συμπεριφορές ιδιαίτερα όσον αφορά την παράνομη ε, απόρριψη επικίνδυνων απορριμμάτων. Αν εγκριθεί λοιπόν η μεταρρύθμιση και αν συσταθεί αυτό το Διεθνές Δικαστήριο θα διευκολυνθεί η δεύτερη μεταρρύθμιση. 20 χώρες της Ένωσης ήδη είναι μεγάλο ποσοστό το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο για το Περιβάλλον θα βοηθήσει στη δράση του άλλου, ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Περιβάλλον. Ιστορικοί λόγοι και μεγάλες καταστροφές που πέρασαν ατιμόρυτες και μεγάλη ζημιά και για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον. Παραδείγματος, τι έγινε μετά τον Ποπάλ, με 30.000 νεκρούς. Περίπου 500 ευρώ πήρε ο κάθε συγγενής θύματος. Ποινικές κυρώσεις το 2010, δηλαδή 26 χρόνια μετά την καταστροφή. Δεν διώχθηκαν οι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και καμία αποκατάσταση για το περιβάλλον. Τελεία απουσία ευθύνης της επιχείρησης. Μία μη δικαιοσύνη ουσιαστικά με δύο λόγια. Αυτό ζήσαμε. Κάτι που είναι σε αντίθεση με τις αρχές της Ένωσης που μιλάει για κυρώσεις αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές. Και ένα απλό ερώτημα στο σημείο εδώ. Αν οι μεγάλες καταστροφές του περιβάλλοντος που είχαμε τα τελευταία χρόνια με καταστροφή των οικοσυστημάτων μπορούν νομικά να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σας θυμίζω εντάχει τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 121, 22, 123. Σας θυμίζω εντάχει το άρθρο 7 το ότι Μιλάμε για ανθρώπινες ενέργειες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια καταστροφή και το περιβάλλοντος έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. χωρίς βέβαια να θέλουμε να περάσουμε σε υπερβολές στη δράση της δικαιοσύνης. Τώρα έχουμε σε μια τρίτη πρόταση μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την τελευταία καταστροφή που το βλέπουμε και στο ίντερνετ παρόλα αυτά καθημερινά. Εξακολουθεί το πετρέλαιο να βγαίνει στη θάλασσα, στον κόλπο του Μεξικού. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται η καταστροφή και βλέπουμε την τεράστια ποσότητα των υδρογοναθράκων που υπολογίζεται. Μπορούμε να δούμε το νούμερο συνεχώς στο Ιντερνετ. Ποια είναι η πρόταση. Πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή, να συσταθεί μια επιτροπή με συγκεκριμένες προδιαγραφές και έργο, επιστημονική βέβαια. Και χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Καταρχήν χρειάζεται τεκμηρίωση. Και όλα αυτά τα στοιχεία να δοθούν στα κράτη-μέγη της Ένωσης που υπέγραψαν στη Ρώμη το καθεστώς του ποινικού αυτού δικαστηρίου για να αποφευχθούν τέτοιου είδου ε, ε, καταστροφές του περιβάλλοντος που γίνονται με σκοπιμότητα και πρέπει να χαρακτηρίζονται ως έγκλημα κατά τη ανθρωπότητας. Υπάρχουν ε, τα άθρα της συνθήκης, υπάρχει προτινόμενη μεταρρύθμιση με περιβαλλοντική καταστροφή εκ προθέσεως. Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο πρέπει να είναι ένα δικαστήριο παράλληλο ως δίδυμο ΟΝ σε σχέση με το Διεθνές Δικαστήριο προτείνεται να υπάρξει μια νομικοεπιστημονική επιτροπή της οποία τα μέλη θα είναι εμπειρογνώμονε με συγκεκριμένους στόχους να συντάξουν το καθεστώ του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαστηρίου τι αρμοδιότητε θα έχει τι νομικά εργαλεία πρόληψης θα διαθέτει και το πιο σημαντικό είναι αυτό, όχι η καταστολή, η πρόληψη ευανομικά εργαλεία καταστολής και πώς θα λειτουργεί. Να τοποθετηθεί αυτό μέσα στο όλο αρχιτεκτόνιμα της Ένωσης με διάσταση προστασίας της υγείας και με σεβασμό και της πολιτιστικής πτυχής. Και τέλος, Υπάρχουν οι αναγκαίε έννοιε για να μπορούν να κρίνονται πότε υπάρξει ρήπανση του περιβάλλοντο, αξιολόγηση τη ζημιά που έγινε στον τοπικό πληθυσμό και στο οικοσύστημα και η ε, καταστροφή περιβάλλοντος εκ προθέσεως που θα χαρακτηρίζεται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτές, σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε και τελειώνω με μερικά σύντομα τηλεγραφικού χαρακτήρα σχόλια. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις που σας ανάφερα, η Διεθνής Ακαδημία ε, Περιβαλλοντικών Επιστημών ελπίζει ότι η Επιτροπή σας θα αξιολογήσει τις προτάσεις μας Είμαστε στη διάθεσή σας να δώσουμε ό,τι πόρους έχουμε προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Η Ακαδημία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής σας την Βίλα Έριον στην Τζουντέκα και στην Αγία Ελένη, στη Βενετία, για το πρόγραμμα για το δικαστήριο και ευχόμαστε η Επιτροπή σας να γράψει μια ιστορική σελίδα σχετικά με την πρόληψη και την καταστολή των περιβαλλοντικών καταστροφών που έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση του ανθρώπου πολύ πριν καταδικαστεί από τον νόμο. Και σας καλώ όποτε θέλετε να κάνετε την επόμενη συνεδρίασή σας στην Βίλα Έριον. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ καθηγητά Αμπράμι για τα όσα μας εξηγήσατε. Γιατί ακούσαμε από το στόμα σας την ε, εξήγηση, την ανάλυση αυτής της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό ποινικό περιβαλλοντικό δικαστήριο. Πάρα πολύ σωστή η πρωτοβουλία σας. διότι το περιβαλλοντικό έγκλημα πολύ συχνά μένει ατιμόρυτο όπως είπατε και αυτό είναι απαράδεκτο. Έχουμε επομένω κάποια ελάσσον εγκλήματα και δηλαδή κάποια πάρα πολύ σημαντικά από αυτό που μας αναφέρατε ε, είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ παραβλάπτει τους φυσικούς πόρους, τις, ε, τους ανθρώπους τελικά, ολόκληρες κοινότητες και πάρα πολύ λίγες είναι οι χώρες οι οποίες ε, έχουν κάποιο πλαίσιο νομοθετικό τόσο ώστε να επιβάλλονται κυρώσεις στους ε, αυτούργους αυτών των εγκλημάτων και εδώ μιλάμε τώρα για κάποια δημόσια αγαθά, ε, υπερσυνοριακά, ε, υπερεθνικά, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, είναι το οικοσύστημα. Και βεβαίως το εθνικό δίκαιο δεν αρκεί. Πάρα πολύ επομένω. Το ότι ήρθατε εδώ και όλα αυτά μα τα εξηγήσατε για να κάνουμε κάτι, να προωθήσουμε αυτή την ιδέα. Άλλωστε έχουμε κάποιου συναδέλφου οι οποίοι έχουν ε, ερωτήσει να υποβάλουν. Πρώτο ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. ευχαριστώ κύριε καθηγητά Αμπράμι για την παρουσίαση που μα κάνατε. Εγώ θα ήθελα να δω το θέμα πολιτικό, επειδή είμαστε πολιτικοί. όχι το στο προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση του πλανήτη σήμερα. Έχουμε μία de facto παγκοσμιοποίηση. Πάμε ξάρει η υπερθέρμανση του πλανήτη. έχουμε το φαινόμενο θερμοκηπίου με τα σχετικά αέρια. Σε οποιοδήποτε σημείο της γης γίνει αυτή η εκπομπή, επηρεάζει όλη την ατμόσφαιρα, σε όλη τη γη. Άγιοι με δύο λόγια. Εδώ χρειάζεται διαχείριση αυτής της αλληλεξάρτησης. Πολιτικά δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ένα σύστημα κυβέρνησης έστω και με μικρή αρμοδιότητα, αλλά πρέπει να υπάρχει. Είναι υποχρεωτικό αυτό το συμπέρασμα. Και πρέπει να κρίνουμε μια έννοια που μέχρι τώρα ήταν θεμελιώδης, δηλαδή την έννοια της εθνικής ή ας το πούμε της επικυριαρχίας. Πρέπει να το ασκήσουμε κριτική. Δηλαδή, Ανέκαθεν ξεκινούσαμε από την κουλτούρα του εθνικού κράτους και λέμε ότι η επικυριαρχία είναι μια απόλυτη έννοια που είναι επαφίεται 100% στο εθνικό κράτος. Ε, λοιπόν, η πολιτική ορίμανση έγκυται σε αυτό. Αυτό δεν είναι αλήθεια πια. Δεν αληθεύει. Για τον το λόγο ότι υπάρχουν στοιχεία που μας δείχνουν ότι ζούμε μια κατάσταση αλληλεξάρτησης. Αν θέλουμε λογικά να δώσουμε μια απάντηση, τίθεται θέμα διακυβέρνησης, κυβέρνησης και δικαιοσύνης. Διαφορετικό. Και θα πρέπει να κινηθούμε στο σωστό επίπεδο Θέλω να επιστήσουμε την ανάγκη να συμπληρωθεί μια άλλη αρχή που είναι η αρχή της επικουρικότητας. που δεν μπορεί να ερμηνεύεται μόνο σε ένα πέρασμα από ένα επίπεδο αρμοδιοτήτων από το πιο ψηλό προς ένα επίπεδο πιο χαμηλό. Η έννοια της υποκουρικότητας πρέπει να λειτουργεί αμφίδρομα. Δηλαδή, τα διεθνή θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο εθνικό. Πρέπει να συμφωνήσουμε για το πώς συνενετικά θα διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Θετικά. Με πολιτική λύση. Και τίθηκε το θέμα και σε ποινικό επίπεδο. Η απόλυτη έννοια της επικυριαρχίας και εδώ παρεμβαίνει. Φερπίνη η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τι λένε, ένας Αμερικάνος πολίτης δεν μπορεί να δικαστεί παρά μόνο από Αμερικανικό δικαστήριο. Ε, είναι σωστό αυτό, κατά τη γνώμη μου, όχι. Υπάρχουν ευθύνε που πάνε πέραν του εθνικού επίπεδου. Φυσικά χρειάζεται πολλή δουλειά για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Αντικειμενικά όμως αυτό οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση, απορρέει από την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία που κατά θα είναι υπερεθνικά. Και εμεί ω Ευρώπη έχουμε εμπειρία από αυτό. Να υπάρξει δηλαδή ένα νέο επίπεδο διοικητικό, υπερεθνικό, που θα μας επιτρέψει να κυβερνούμε σε σχέση με τα προβλήματα αυτά που είναι υπερεθνικά. Στην Ευρώπη ήδη έχουμε κάνει βήματα, αλλά κάπως δειλά. Στόχος θα είναι να βρεθεί μια λύση και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για το περιβάλλον. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε Βικτόριο για τη βαθιά αυτή φιλοσοφική ανάλυση. Εύστοχη παρέμβαση. Γιατί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην υπερεθνικότητα και στην επικουρικότητα. Στην εθνική επικυριαρχία και των υπερεθνικών εγκλημάτων που διαπράττονται κατά το περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον δόκτωρα Αμπράμι για την παρουσίαση αυτής του της ε, πρωτοβουλίας αν κανείς θέλει να είναι αισιόδοξο, θα πρέπει να παραδεχθεί ότι έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα σχέση με το περιβάλλον και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε να έχουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Βέβαια καταλαβαίνω ότι τώρα απλώς έχουμε έναν καταιγισμό ιδεών, όπως λέμε, και να δούμε τώρα κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα πρώτα-πρώτα. Τι αρμοδιότητα, τι ειδικία θα έχει αυτό το δικαστήριο ανακριτικές ενέργειες, επιβολή κυρώσεων. Τι, τι, τι θα μπορεί να κάνει πιο συγκεκριμένα. Να κάτσουμε και να δούμε το ότι αυτό το δικαστήριο θα δικάζει ποιον. Θα μπορεί να εγκαλέσει εκεί νομικά πρόσωπα ή και φυσικά πρόσωπα. Φυσικά και ο τόπος εγκαταστάσεως του δικαστήριου είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε την τραγωδία του Γκολ του Μεξικού. Είδαμε εκεί ότι μια εταιρεία είναι ο υπεύθυνο. Σε κάποιε άλλε περιπτώσει, όπω στην περίπτωση τη Βαλτική θάλασσα, έχουμε περισσότερε φορεί, περισσότερα μικρά πρόσωπα τα οποία ευθύνονται για την αυξανόμενη τοξικότητα τη θάλασσα εκείνη. Καμιά φορά έχουμε δραστηριότητε κάποιων ε, εταιρεών που όντως προκαλούν μόλυνση. Αλλά δεν είναι μετρήσιμη η μόλυνση αυτή, η ευθύνη αυτή. Αν θέλουμε ένα ενωσιακό, ένα δικαστήριο για την ΙΟΚ, μήπως τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί είναι πιο προχωρημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα θέματα τα νομικά και τα δικαστικά. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλουμε να καλύψουμε και τρίτες χώρες όπως την Κίνα, την Ρωσία ή την ε, ΙΠΑ ή την Λευκο-Ρωσία ε, τι θα γίνει. Äh, Ευχαριστώ, Νικ Γκρίφιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον ε, καθηγητή για την τόσο συναρπαστική του εισήγηση. Για πέστε μου, η Ακαδημία σας είναι υπέρ του να χρησιμοποιηθεί αυτό το δικαστήριο για να κάνουμε κάτι, να καταπολεμήσουμε αυτή την προπαγάνδα, να εγκαλέσουμε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την υπερθέμιση του πλανήτη. Πρόεδρος. Πάρα πολύ προκλητική ερώτησή σας. Και τώρα έχουμε τη Γιολάντα Φίπνερ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Αβράμη. Πολύ ωραία πρωτοβουλία να υπάρξει αυτή η μονάδα ελέγχου, το όργανο ελέγχου. Ιδιαίτερα μάλιστα αν μπορεί να δράσει σε διεθνές επίπεδο. Η σύσταση ενός τέτοιου οργάνου όμως θα, θα, θα κρίνει και τα αποτελέσματα των καταστροφών αυτών, των οικολογικών καταστροφών. Από ό,τι κατάλαβα, μιλήσατε και για ένα σύστημα κυρώσεων ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής. Στον τύπο αυτή τη στιγμή διαβάζουμε ότι η BP δεν έλαβε υπόψη αυτό που έλεγαν οι ειδικοί για το πόσο επικίνδυνο ήταν το εξορρυκτικό της εγχείρημα στις δικές σας πρωτοβουλίες προβλέπετε και μία συνεργασία με τα ελεγκτικά όργανα, διότι ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε το πρόβλημα αφού έχει γίνει η ζημιά, αλλά και η πρόληψη είναι σημαντική. Ερωτώ λοιπόν τον καθηγητή, προβλέπονται συστήματα προληπτικού ελέγχου, πρόληψης, πληροφόρησης ή ένα σύστημα προληπτικών κυρώσεων για να μην καταλήξουμε στην οικολογική καταστροφή Πρόεδρος. Και συνάδελφος Λίχτενμπεργκερ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι επισκέπτρια από την Νομική Επιτροπή όπου ήδη ασχοληθήκαμε με κλίμα κατά του περιβάλλοντος διασυνοριακά, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα de facto. Δεν είναι σύμπτωση τότε ορισμένες επικίνδυνες μονάδες πολύ συχνά είναι κοντά στα σύνορα από τεφροτήρες, από ρημάτων, πυρηνική σταθμή, ε, μονάδες που ρίχνουν επικίνδυνα υλικά στα ποτάμια είναι πάντα κοντά στα σύνορα, πολύ συχνά μάλλον. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως εμένα ιδιαίτερα είναι αν, αν υπάρξει ένα τέτοιο ευρωπαϊκό ή διεθνές δικαστήριο πώς θα, τι νομική βάση θα πρέπει να του δώσουμε έτσι ώστε πραγματικά να είναι δεσμευτικό στη δράση του για τα κράτη-μέλη, μιλάω τώρα για την Ευρώπη, όπου να έχει ε, ποινική ισχύ σε θέματα ζωής και θανάτου. Γιατί στην Νομική Επιτροπή είχαμε μερικές παρόμοιες περιπτώσεις κρούσματα, εγκλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα και το θέμα είναι πρέπει να υπάρχουν ποινικέ κυρώσει. Είπαμε εμεί και το Συμβούλιο μέχρι στιγμής όλα αυτά τα μπλοκάρει και τα απορρίπτει. Είμαστε μένει στην Ένωση, αλλά ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στο δρόμο αυτό ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας δράσης όταν επισυμβαίνει κάτι διασυνοριακά. Το έχετε σκεφτεί αυτό, τι ενδεχόμενες λύσεις, πώς θα μπορούσαμε να κινήσουμε τη διαδικασία αυτή. Ε? Γιατί ο δρόμος αυτός είναι πολύ πιο δύσβατος από ό,τι φανταζόμαστε. Και αν άρουμε μερικά από τα μικρά εμπόδια που υπάρχουν στο δρόμο αυτό, και αυτό από μόνο του καλό είναι. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου εκ μέρου της Νομική Επιτροπή. Τη χρειαζόμαστε. Μέχρι στιγμή ε, το ποινικό δικαστήριο, το ποινικό δίκαιο αναφέρεται σε θέματα ζωή και θανάτου ή κινδύνου τη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Οπότε εδώ χρειαζόμαστε, επειδή μιλάμε για το περιβάλλον, χρειαζόμαστε νέες βάσεις, νέα στοιχεία. Από ό,τι κατάλαβα, η συνθήκη της Ρώμης, που αποτελεί και τη βάση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα κατά της ανθρωπότητας, πρέπει να διευρυνθεί αυτή η σύμβαση της Ρώμης. για να συμπεριλάβει το οικοσύστημα και ως εκ τούτου να αποτελέσει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ή καταστροφή του οικοσυστήματος. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει η αναλογικότητα και στο εθνικό σύστημα. Θα υπάρχει δυνατότητα ανάληψης δράσης. Δηλαδή, και εφόσον δεν προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο από την νομοθεσία η ποινική διαδικασία, τότε θα μπορεί να λαμβάνει το διεθνές ποινικό δικαστήριο. Το ευρωπαϊκό τώρα τι θέση θα έχει. θα έχει κάποιο λόγο ύπαρξης ή όχι. Μια σειρά ερωτήσεων λοιπόν για τον κύριο Αβράμι. Και η Κάριν Κάρενμπαχ. Πολύ σύντομα για διευκρίνηση. Ναι και δεν είμαι νομικός. Μόνο για ποινικά ζητήματα θα είναι αρμόδιο το δικαστήριο αυτό έτσι δεν είναι το το ποινικό όμως ε, αδίκημα προϋποθέτει είτε αμέλεια βαριά ή δόλο. Εάν δεν υπάρχει αμέλεια ή δόλος δεν θα καλύπτονται προφανώς αυτά τα προβλήματα από την ε, δικαιοδοσία του ποινικού δικαστηρίου. Μένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιο κάνει τον προσδιορισμό, γιατί έχουμε σαφεί προσδιορισμού τη νομική βάση για άλλα εγκλήματα, αλλά όχι για τα εγκλήματα ει βάρο του οικοσυστήματο. Ο πρόεδρο αφαιρεί τα ερωτήματα, τώρα έχετε και την ευκαιρία να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ του ε, ευρωβουλευτέ. Οι ερωτήσει σα ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντικέ. Ας αρχίσω από αυτά που είπε ο καθηγητής Πρόντι. Θέτεται το πρόβλημα της εφαρμογής κυρώσεων, το πρόβλημα της επικουρικότητας και της ενδεχόμενης παραβίασης της αρχής επικυριαρχίας. Σπέβδω να δηλώσω ότι στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του ποινικού δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού με αυτά δεν παραβιάζεται η αρχή της επικυριαρχίας. Γιατί όλοι ξέρουμε να πάρουμε το Ιταλικό Σύνταγμα αλλά και τα άλλα συντάγματα ισχύει αυτό ότι το, το ποινικό πεδίο κάθε κράτος ζηλότυπα κρατάει την επικυριαρχία του και ορίζει αυτό τις ποινές και τις κυρώσεις για συμπεριφορές που αποτελούν αδίκημα ή έγκλημα. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη μεταρρύθμιση και το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο Περιβάλλοντος. Γιατί? Διότι κάθε χώρα της Ένωσης θα συνεχίσει να έχει το δικό του ποινικό δίκαιο. Θα οφείλει να εξασφαλίσει μια ομοιομορφία με βάση την οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου με κυρώσεις που θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες σε σχέση με άλλες ποινές που επιβάλλονται για παρόμοιες περιπτώσεις και συμπεριφορές εγκληματικού χαρακτήρα στις άλλες χώρες. Άρα κάθε χώρα θα εξακολουθεί να ορίζει τα εγκλήματα πότε μια συμπεριφορά αποτελεί έγκλημα ή αδίκημα με βάση αυτό που θα έχει ορίσει η Ένωση μέσω της οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Και από εν μέρη σε μια άλλη ερώτηση, σε σχέση με το θέμα της ε, υπερθέρμανσης του πλανήτη. γιατί τιμωρούνται συμπεριφορές από την εμπορία προϊόντων που επηρεάζουν, παραδείγματος χάρη, το στρωματόζοντος. Σε τι συνίσταται τώρα και στο σημείο αυτό πολύ σωστά είπε αυτά που είπε ο καθηγητής Πρόντιο και οι άλλοι ευρωβουλευτές βέβαια, από άλλη πλευρά όμως όταν αναφέρθηκε στην αρχή της επικορικότητας, διότι με την αρχή της επικορικότητας ακριβώς υλοποιείται η σύσταση του ποινικού δικαστηρίου. Γιατί ο πρόεδρος πριν ανάφερε το σύστημα το ποινικό δικαστήριο παρεμβαίνει εκεί που δεν παρεμβαίνει ο εθνικός δικαστής. Δεν υποκαθιστά τον εθνικό δικαστή. Έχουμε ενοποίηση των συστημάτων. Έχουμε δηλαδή μια διαδικασία εξισορρόπησης και αντιστάθμισης. Ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε τη Ρουμανία και τα Ορουλ τι θα είχε γίνει αν είχαμε Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο και να έχουν ρίξει 100.000 κυβικά μέτρα τοξικής ύλης στο ποτάμι. Κάτι θα είχε γίνει. Θα είχε γίνει ότι ο Πέτρος, επί του περιβάλλοντος δεν θα κατέληγε στο συμπέρασμα που κατέληξε τα χέρια ψηλά, δεν υπάρχει προστασία. Αυτό σίγουρα μπορούμε να το πούμε και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Όχι παραβίαση λοιπόν του ποινικού δικαίου εθνικά. Η κάθε χώρα μπορεί και θα οφείλει να εντοπίσει με ποιες κυρώσεις θα κινηθεί κατά των πράξεων αυτών. Άλλο πράγμα όμως, η πρόβλεψη των ποινών και άλλο η επιβολή των ποινών. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό σας είπα αποτελεσματική δικαιοσύνη. Η Ένωση εδώ και χρόνια μιλάει για την αναλογικότητα των ποινών, την αποτρεπτικότητα των ποινών. Τι αποτρεπτικότητα υπάρχει όμως όταν δεν εφαρμόζεται η ποινή, μένει στα χαρτιά. Υπάρχει λοιπόν δημιουργείται ένα κίνητρο Σωστά αναφέρθηκε το ότι το ποινικό δικαστήριο, το διεθνές δικαστήριο που υπάρχει, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν συμμετέχουν σε αυτό το δικαστήριο. Δεν θα δεχτούν ποτέ, λέτε, οι Ηνωμένε Πολιτείες αν έχουμε, ας πούμε, ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο για το περιβάλλον να, να γίνουν μέλος αυτού του δικαστηρίου. Ζηλότυπα θα κρατήσουν την επικυριαρχία τους. Κύριε καθηγητά Πρόντι, εγώ θεωρώ ότι αν εμείς το 1972, όταν είχαμε την πρώτη διεθνή διάσκεψη στη Στοκχόλμη, αν δεν είχαμε προβλέψει ότι μετά από 20 χρόνια θα γινόταν αυτά που έγινε για το περιβάλλον, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη για το θέμα του περιβάλλοντος στις συνειδήσεις των ανθρώπων όπως έγινε. Δηλαδή, αν είχαμε προβλέψει ένα Ινστιτούτο πρόληψης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την αρχή Μπράτλαντ ποτέ δεν θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Γι' αυτό σας είπα ότι είμαι αισιόδοξο. Μια δεύτερη ερώτηση, ποια είναι είναι η λειτουργία του ποινικού δικαστηριού. Ποιος θα είναι ο ρόλος λοιπόν, κυρίως προληπτικός. σκεφτείτε ένα, ένα που μπαίνει στα χωρικά είδετα της Ένωσης ένα, με επικίνδυνο φορτίο. Πριν γίνει η καταστροφή, εγώ ως δικαστής μπορώ να το κατάσχω το πλοίο αυτό, να κατάσχω το φορτίο του. Αν δεν το κάνω εγώ, ο Ευρωπαίος δικαστής, μπορεί να το κάνει ο Εθνικός Δικαστής. Αν δεν το κάνει ο Εθνικός Δικαστής, μπορώ εγώ ως ποινικό δικαστήριο να παρέμβω. νομικό, νομικά χαρακτηριστικά, αν υπάρχουν εξουσίες που δεν ασκούνται, η σχέση των ποινών σε σχέση με τη ζημιά κλπ. Αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά οι βασικές νομικές αρχές νομίζω είναι σαφές. Βαλτική θάλασσα, ρήπανση, πώς θεωρίζονται οι ευθύνε κλπ. Κοιτάξτε, με βάση αυτό είναι δυνατόν να προβλεφθεί. Το θέμα, το θέμα της ζημιάς στο περιβάλλον είναι το πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι καθοριστικό. Και δεν είναι μόνο η οικολογική ζημιά, όπως είπα και πριν, είναι και η βιολογική ζημιά. Οι ανθρώπινε σχέσει δοκιμάζονται. Όλα αυτά πλήττονται από μια οικολογική καταστροφή. Ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ και τον Δ. Κρόνοτ και τον καθηγητή τον Ρομπέρτο Ταντόνι που ήρθαν. Τι Ρομπέρτο Ταντόνι. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Και η προσπάθειά σας, τα όσα είχατε να μας πείτε. Σημειώνουμε λοιπόν την πρωτοβουλία σας. Υπάρχει πολύ υλικό ακόμα να διαβάσουμε. Νομίζω ότι δώσατε τροφή για συζήτηση, για σκέψη και θα πρέπει νομίζω να προχωρήσουμε και να κλείσουμε τα κενά. στον έχουμε ένα μηχανισμό κυρώσεων για την ε, αναγνώριση των ευθυνών και την επιβολή κυρώσεων ποινικών, ενδεχομένως προληπτικά ως προς τα αγαθά του περιβάλλοντος και τα οικοσυστήματα. Κυρίε και κύριοι, ολοκληρώνεται τη συνεδρίασή μας. Όποιος λοιπόν δεν έχει ε, την πρόθεση να συμμετάσχει στη συνεδρία των συντονιστών, μπορεί να αποχωρήσει. Σας εύχομαι καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση 6 Σεπτεμβρίου. Αυτά το απόγευμα σε ειδική συνεδρία στο Στρασβούργο. Θα τα ξαναπούμε. Πέρα στη σου. συντονιστέ. Χαίρετε. Okay.